από την ομάδα S&D έλαβα κάποια αιτήματα τροποποίησης ε, στους ε, ορισμούς επιτροπές και σε αντιπροσωπίες. Αυτά θα δεγραφούν στα πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης. Αν δεν υπάρχουν παρατηρήσεις μέχρι την έγκριση των πρακτικών, θα